witam państwa ponownie. Αρχίζει πάλι η συνεδρίαση. Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση του κυρίου Φλέκενστάιν για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων. Συγγνώμη. Ο κύριος ε, Φλέκενστάιν προέρχεται από μια πόλη λιμάνι. Του δίνω λοιπόν αμέσω το λόγο. Κύριε Φλέκενστάιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, από την αρχή της συζήτησης για το πακέτο λιμένων